Ε, ε, αυτό το κοινοβούλιο διότι ήταν δύσκολο για μένα φυσικά να παρακολουθώ την αποχώρηση, της, ε, την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου ως Ιρλανδός λόγω των δεσμών που έχουμε με τη χώρα αυτή. Όμως βρισκόμαστε σε μια πολύ διαφορετική κατάσταση είναι πραγματικά ε, λυπηρό το ότι μιλώ πρώτη φορά εδώ για το Brexit γιατί αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο κατέβηκα στην πολιτική πριν από ένα χρόνο και τελικά υπό περίεργες συνθήκες βρέθηκα εδώ. Βρισκόμαστε σε ένα λεπτό σημείο των διαπραγματεύσεων ε, της διαδικασίας αυτής και δεν υπάρχει ε, ιστορικό προηγούμενο ε, ε, εμπορικοί εταίροι να προσπαθούν να καθορίσουν εμπορικά εμπόδια. Οπότε θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη μας ε, την, το γεγονός ότι οι Βρετανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την έκπληξή τους όσον αφορά την φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλλει κανόνες στο, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λαμβανωμένου υπόψη ότι και οι Βρετανοί οι ίδιοι συνδιαμόρφωσαν αυτό το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι ε, θα πρέπει να προσεγγίσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο ως μελλοντικό εταίρο και συνεργάτη και όχι να το τιμωρήσουμε για την αποχώρησή του. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βιλίμσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία το, το, το, το γεγονός ότι δεν έχουμε πια μαζί μας τους ε, Βρετανούς για να ε, ευχηθώ και να συγχαρώ τους Βρετανούς για την ε, νέα τους ανεξαρτησία και ότι το έχουν αποδεσμευτεί πλέον από το κέντρο λήψης αποφάσεων των Βρυξελών και ότι πλέον το κέντρο λήψης αποφάσεων θα είναι το Λονδίνο. Σε κάποιους μπορεί αυτό να αρέσει και σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει. Πάντως γεγονός είναι ότι όλα αυτά έγιναν ε, έπειτα από ένα δημοκρατικό δημοψήφισμα και παρόλο που προσπάθη, επιχειρήθηκε από διάφορες πλευρές να αναγκαστούν οι Βρετανοί να παραμείνουν παραμείνουν με διάφορα τρίκ στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Βρετανοί οι ίδιοι ε, απέδειξαν ότι η πλειοψηφία ήταν υπέρ του Brexit. Και τώρα εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να προσεγγίσει τους Βρετανούς με αυτή τη νέα τους ανεξαρτησία, με φιλικές σχέσεις, με ευελιξία ή θέλουμε να τους κακομεταχειριστούμε και πάλι με την επιβολή κανόνων από τη δική μας πλευρά ή να τους ε, καταδιώξουμε, να τους διώξουμε ε, σε μια θέση ε, που θα τους οδηγήσει περισσότερο σε μια ατλαντική σχέση. Υπάρχει αυτό το δίλημα μπροστά μας. Θέλουμε να είμαστε φιλικοί και ευγενεί απέναντί τους ή θέλουμε απλά να τους διώξουμε από κοντά μας. Ευχαριστώ. Επόμενη, επόμενη, επόμενη ο κύριος Φερέιρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συζητάμε τι μελλοντικέ σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένου Βασιλείου. Μα προφανώ οι σχέσει αυτέ θα έχουν να κάνουν με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αυτών. Εμεί θέλουμε να προωθήσουμε συγκεκριμένε ισχυρέ θέσει όσον αφορά τα περιβαλλοντικά κοινωνικά μα πρότυπα όσον αφορά την οικονομία μας, όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων. Έχουμε άραγε αντίστοιχη στάση από το Μένο Βασίλειο ή μήπω βλέπουμε εκεί πέρα μια πιο επιθετική στάση ακόμα και στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου και των εξωτερικών πολιτικών. Μια μηδέα εποφελής πολιτική χρειάζεται και σε άλλους τομείς όπως ο πολιτισμός. Χρειαζόμαστε εδώ πέρα να έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας όπου θα διασφαλίζεται η κυριαρχία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Μένο Βασιλείου προ το όφελο όμως των πολιτών και στις δύο πλευρές της μάχης, σε καμία περίπτωση εις βάρος τους. Οποιεσδήποτε και είναι οι περιστάσεις, δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσουν σε εκχωρήσεις οι οποίες τελικά θα είναι επιζήμιες για τους πολίτες τους και δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι η μόνη η οποία θα αποφασίζει για τις διαπραγματεύσεις αυτές τη στιγμή που ξέρουμε ότι το Μένο Βασίλειο θέλει και αυτό να έχει συγκεκριμένο λόγο όσον αφορά την απελευθέρωση του εμπορίου. Ο κύριος Μουρεσάν έχει το λόγο. Κύριε Μπαρνιέ, είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε την ενότητα των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Brexit διέρεσε για πάρα πολλά χρόνια τον πληθυσμό της, του Ηνωμένου Βασιλείου. Το ίδιο έγινε και με τη Βρετανική κυβέρνηση και οδήγησε σε πρόορες εκλογές. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως εμείς επιτελέσαμε την εντολή μας, καταφέραμε με εντελώ αποτελεσματικό μη τρόπο να κάνουμε σωστά το δικό μα το έργο και να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου από όλε τι πολιτικέ ομάδε. Τι θέλουμε τώρα να πετύχουμε. Πρώτη προτεραιότητα. Δικαιώματα των πολιτών. Βεβαιότητα για του αγρότε, του ερευνητέ, του φοιτητέ σε σχέση με τη μελλοντική αυτή σχέση. Ο στόχο μα θα πρέπει να είναι μια σχέση ω τον πιο στενή με τον Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα όμω τα μέσα είναι απόλυτα ξεκάθαρα. Μια σχέση που θα βασίζεται σε κανόνε. Είναι πολύ σημαντικό να τηρούνται σε κάθε περίπτωση οι κανόνε. Και θα πρέπει οποιοδήποτε αποτέλεσμα έχει η διαπραγματευτική και αυτή εντολή να ευθυγραμμίστε με τις προθέσεις και τους στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπω περιγράφονται στο ψήφισμα αυτό. Ευχαριστώ. Η επόμενη μιλήτρια είναι η κυρία Ίνσιρ. Κυρία Πρόεδρε, το Brexit είναι ένα θλιβερό κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή ιστορία. Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία και όχι λιγότερη. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε σταθερότητα και ελευθερία στην Ήπειρό μας. Μια Ήπειρος η οποία έχει πληγεί από συγκρούσεις και πολέμους στην ιστορία της. Τώρα οι εθνικιστικές δυνάμεις στην Βρετανία κατάφεραν και πραγματοποίησαν το όνειρό τους. Όμως είναι σημαντικό παρόλα αυτά να μπορέσουμε να συνάψουμε μια καλή συμφωνία με τους Βρετανούς. Πρέπει να υπερασπιστούμε τις κατακτήσεις της ενιαίας αγοράς, την, ε, το ευρωπαϊκό δίκαιο που έχουμε οικοδομήσει, τα φιλόδοξα πρότυπά μας όσον αφορά την περιβαλλοντική και κοινωνική πολιτική. Ο κύριος Τζόνσον δεν μπορεί να φύγει νικητής ε, από όλη αυτή τη διαπραγμάτευση. Τα ψέματά του αρκετό κακό έχουν ήδη προκαλέσει. Γι' αυτό και πρέπει με ενιαίο τρόπο, με ενότητα να εμφανιστούμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Θέλω να πω στους νέους της Βρετανίας, μην τα παρατάτε. Υπάρχουν πάρα πολλοί εδώ μέσα που έχουν το, μέλλον, το, το βλέμμα του στραμμένο στο μέλλον και νομίζω ότι οι δρόμοι μας μπορούν να ξανασυναντηθούν. Ε, κύριε Νετφέλτ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε σκληρή γλώσσα για την εξασφάλιση ισότιμων κανόνων παιχνιδιών και ότι δεν θα ρίξουμε τις προδιαγραφές μας, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των τροφίμων ή τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Ελπίζω οι διαπραγματευτές να είναι εξίσου σκληροί όταν πρόκειται για τα πρότυπα προστασίας των προσωπικών δεδομένων διότι αγωνιά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λύσει το θέμα της ε, απόφασης καταλληλότητας, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να χειρίζεται ε, τα δεδομένα μας με τρόπο ε, σωστό. Και αναφέρομαι στο πρόσφατο σκάνδαλο με την πρόσβαση στην Τράπεζα Δεδομένων του Σέγγεν του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι ιδιαίτερα τα δικαιώματα των πολιτών και ε, απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντονότατη. Είναι 3,5 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ε, πολίτες ε, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1,5 εκατομμύριο Βρετανοί στην Ευρώπη των 27. Και παρακαλώ να βεβαιωθείτε ότι αυτά θα είναι εγγυημένα όχι μόνο στα λόγια αλλά και στα έργα. Ο κύριος Μπούχαϊτ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, εδώ στην Ολομέλεια θεωρούμε εκπρόσωπος μιας κοινότητας που κινδυνολογεί, ε, που υποδαβλίζει συναισθήματα βάσιμα. Εμείς δεν είπαμε τίποτα για τα φάρμακα και για τα τρόφιμα που θα ε, ε, σπάνιζαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τον Brexit ή θα είχαμε κυκλοφοριακό χάος ε, στα σύνορα. Δεν τα λέμε εμείς αυτά. Οι εκπρόσωποι του λεγόμενου αστικού κέντρου. Ε, σήμερα ποια είναι η δυσκολία ότι δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε μια δημοκρατική απόφαση του λαού. Δεχτείτε ως συνομιλητή ε, ισότιμο το Ηνωμένο Βασίλειο και τώρα σκεφτείτε και κοιτάξτε τις νέες δυνατότητες ως μια νέα αρχή, ως μιας δυνατότητας να φτιάξουμε γέφυρες παρά να συνεχίζουμε εδώ με σκληρά λόγια και σκληρά για τις σχέσεις μας και από αυτή την πλευρά της μάχης και από την απέναντι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέλαμι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η σχέση που θα οικοδομηθεί ανάμεσα στις δικές μας χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι αποφασιστική σε πάρα πολλούς τομείς. Υπόθηκαν ήδη πολλά σημαντικά. Θέλω να επανέλθω σε ένα ε, βασικότατο που είναι το ζήτημα της αλίας. Γνωρίζουμε ότι ε, η αλία κυριάρχησε και καθόρισε τον Brexit ε, στη Βρετανία. Σήμερα μόνο χαμένοι θα βγούμε εάν η αλία βγει από τη συνολική διαπραγμάτευση με τους Βρετανούς. Και ε, χαίρομαι, ε, είμαι πολύ ικανοποιημένος που ε, από την αποφασιστική δράση του Μισελ Μπαρνιέ έχει ενταχθεί και η Αλία σε αυτή τη διαπραγματευτική εντολή έτσι ώστε να διαπραγματευτούμε μια συνολική συμφωνία μαζί με την Αλία. Θα είναι πολύ ισχυρέ οι εντάσεις στη θάλασσα και μεγάλη οικονομική καταστροφή αν δεν γίνει κάτι τέτοιο και οικολογική. Χρειαζόμαστε κοινή αλλιευτική πολιτική για να διαφυλάξουμε τα είδη των αλλιευμάτων. Και αυτό είναι πάρα πολύ πολύ σημαντικό για το μέλλον των χωρών μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαλντεμόζε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στόχος της διαπραγμάτευσης αυτής με το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι να πρέπει να έχουμε μια φιλόδοξη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ανάμεσα σε δύο σημαντικούς εταίρους, Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτός είναι ο στόχος μας και θεωρώ ότι αυτό είναι σαφές για όλους. Από την άλλη όμω θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφεί και σε κάτι άλλο, στα αιτήματα τα οποία θα προβάλλουμε προ το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να κάνουμε εκχωρήσει όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντο. Σε καμία περίπτωση θα πρέπει να κάνουμε υποχωρήσει στο φορολογικό καθεστώς ή στι κρατικέ ενισχύσει. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφεί όταν λέμε ότι θέλουμε ισοτιμία στη σχέση ανταγωνισμού, ότι θέλουμε ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Βέβαια, τούτων λεχθέντων είναι προ το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήξει σε μια συμφωνία τελικά. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει αυτή τη στιγμή να απογοητευόμαστε από το ότι το Brexit έλαβε χώρα. Α βρούμε καλύτερα κάποιε θετικέ λύσει σε συγκεκριμένου τομεί. Στην Αλία, για παράδειγμα, θα πρέπει να μπορούν να έχουν οι Ευρωπαίοι αλλοί πρόσβαση ισότιμη στα Βρετανικά είδατα. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ράνχελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Η Κροατική Προεδρία, αγαπητοί εκπρόσωποι της Κροατικής Προεδρίας, κύριε Μπαρνιέ, θέλω να υπογραμμίσω δύο διαστάσεις που ενδεχομένως δεν έχουν τονιστεί επαρκώς. Η πρώτη διάσταση είναι το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό υπό ποιε προϋποθέσεις ε, θα ρυθμιστούν τα ζητήματα ασφαλείας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βελσιλίου. Σκεφτείτε μόνο τι τρομοκρατικέ επιθέσει. Η αστυνομική συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών αρχών των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ύψη τη σημασία. Γιατί δεν είναι δυνατόν να μην μπορέσουμε να βρούμε μια συμφωνία σε αυτού του ε, τομεί, στι δύο πλευρέ τη μάχη. Ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έργο να επεκταθεί και στην άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Είναι πολύ εύκολο Κοιτάζοντα τα πράγματα, να διαπιστώσει κανεί ότι η στάση της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πολύ πιο κοντινή σε εκείνη τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση από ότι σε άλλε χώρε. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρξει συνεργασία και στον τομέα τη άμυνα και τη εξωτερική πολιτική. Ευχαριστώ. Η... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Μπαρνιέ, αποδειχθήκατε πολύ καλός διαπραγματευτής και είμαι βέβαια ότι θα καταλήξετε σε σπουδαία συμφωνία. Αυτό που χρειαζόμαστε πρώτα απ' όλα είναι να υπάρξει συμφωνία. Όπως είπε ο συνάδελφο Χουάν Φερνάντο Λόπεθ Αγγιλάρ. Χρειαζόμαστε μια συμφωνία για να μην υπάρξει πρόβλημα. Αλλά αυτή η συμφωνία θα πρέπει να είναι φιλόδοξη και να εκπροσωπεί τα συμφέροντα του αγροδιατροφικού τομέα με τις, ποιότητες, ε, τις ποιοτικές προδιαγραφές που πολύ καλά γνωρίζει το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Αλία, αναφέρθηκαν σε αυτή και πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Είναι πολύ σημαντική. Τα γνωρίζετε πολύ καλά. Έχετε ασχοληθεί με το θέμα αυτό ως Υπουργό Αλία στη Γαλλία, κύριε Μπαρνιέ. Είναι σημαντικό να συνάψουμε συμφωνία πριν την 1η Ιουλίου για να ξέρουμε αν θα μπορούμε να μοιράσουμε σωστά τα μέγιστα επιτρεπτά αλλιεύματα και τις ποσοστώσεις και να μην τα πληρώσει η Αλία τα σπασμένα. Και θα πρέπει να διασφαλιστεί το γεγονός ότι θα έχει λόγο η Ισπανία σε οτιδήποτε συζητάτε για το Γιβραλτάρ. Ευχαριστώ, Νίντερ Μάιερ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώ επίση και τον κύριο Μπαρνιέ, καθώ επίση και όλη την ομάδα που συνέταξε το σχέδιο ψηφίσματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι πολύ θετικό και πολύ θετική είναι επίση και η συζήτηση. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι έχουν πει τα περισσότερα πράγματα, να τονίσω και εγώ κάποια ζητήματα ελεύθερος ανταγωνισμός αλλά και ισότιμος θεμητός ανταγωνισμός. Αυτά τα δύο πάνε μαζί, δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Βάσει των αρχών αυτών μπορούμε να δημιουργήσουμε μια εισβάθος συμφωνία, ευρεία συμφωνία με το Μένο Βασίλειο. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, αλλά ενδεχομένως να μην γίνει αυτό στην πράξη. Υπάρχουν δύο βασικοί περιορισμοί. Πρώτον, πάρα πολλές κόκκινες γραμμές και δεύτερον, πολύ λίγο χρόνο. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι θα πρέπει να καταβάλουμε άοκνε προσπάθειε. Δύο βασικέ αρχέ θα πρέπει να μα κατευθύνουν. Πρώτον, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να υποχωρήσουμε σε σχέση με τι αρχέ μα. Είναι πάρα πολύ σημαντικέ για μα και για του εταίρου μα. Και δεύτερον, αυτό το οποίο είπε το Συμβούλιο. Πιέζει πάρα πολύ ο χρόνο. Πρέπει να είμαστε γρήγοροι, να δείξουμε ευελιξία για να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για όλου του Ευρωπαίου. Σα ευχαριστώ. Ο κύριος Ντάγκελσον τώρα έχει το λόγο από το μάτι Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό οι διαπραγματεύσεις αυτές να χαρακτηριστούν από σαφείς κατευθυντήρες γραμμές. Εμείς διαπραγματευόμαστε ως ενώσεις. Δεν μπορούν ταυτόχρονα να γίνονται και διμερείς ε, διαπραγματεύσεις μεταξύ κρατών μελών και του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης, μιλάμε για ένα ζήτημα ε, που, έχει, ε, που ε, έχει σχέση με την πρόσβαση στην τεράστια ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε, εργασιακά, δικαιώματα, κοινωνικά πρότυπα, περιβαλλοντικά πρότυπα. Αυτά τα ζητήματα έχουν ε, ιδιαίτερη σημασία και στον τομέα των, μεταφορών, των μεταφορών. Διότι αν δεν καταφέρουμε να βρούμε συμφωνία και υπάρξουν εμπόδια στις μεταφορές, αυτό θα ήταν μια καταστροφή το Ηνωμένο Βασίλειο έπαψε πλέον να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό και θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες όσον αφορά την διέλευση, τη διαμετακόμιση προϊόντων από και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Λονδίνου. Εκεί θα πρέπει πάντοτε να τηρούνται και οι ε, ευρωπαϊκοί κανόνες. Ευχαριστώ ο κύριο Πέτερ. Αξιότιμη Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι, το Brexit είναι γεγονό. Το επόμενο βήμα τώρα είναι μια συμφωνία σύνδεση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Βρετανική κυβέρνηση θέλει να κλείσει αυτή τη συμφωνία σε μόλι οκτώ μήνε. Και να μην υπάρξει σκληρό Brexit όμω, γιατί στο Βέλγιο θα χαθούν 42.000 θέσει εργασία. Θα πρέπει να κλείσουμε μια συμφωνία που θα ισχύει από την 1η Πρώτου του 2021. Αλλά Ας μην γελιόμαστε. Μέσα σε 8 μήνες να συνάψουμε πλήρη συμφωνία σύνδεση είναι σχεδόν ανέφικτο. Γι' αυτό θα πρέπει να τολμήσουμε να βάλουμε προτεραιότητε. Πρώτον, οι ψαράδες μας να συνεχίσουν να ψαρεύουν σε βρετανικά ύδατα. Δεύτερον, να υπάρχει ε, ισότιμο ανταγωνισμός για ε, τα ε, κλωστοϊφαντοργικά, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα τρόφιμα και που πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα. Επίσης, συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη. Είναι κοντινός μας γείτονας και θα παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μιγιάν Μον, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να αναφερθώ σε ένα θέμα πολύ σημαντικό που είναι η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου και ιδιαίτερα η Αλία ε, ε, η συνέχιση της αμοιβαία πρόσβασης στα αλλιευτικά πεδία και τα ύδατα. Τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο κύριος Μπαρνιέ αυτά. Θεωρώ εκ των όνου κάνεφο, όπως είπαν και άλλοι, οι Ευρωπαίοι αλληλείς να διατηρήσουν την πρόσβασή τους σε πόρους και ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι πολλά ε, σημαντικά τα μέρη ε, που θίγονται πάρα πολύ αλλιευτικές κοινότητες στην Ένωση και δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές είναι μεγαλύτερη αγορά για τα αλλιευτικά προϊόντα των Βρετανών αλλιέων. Λοιπόν, είναι αμοιβαίο το συμφέρον και συμπληρωματικό. Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα το εξή. Θα πρέπει να είμαστε στεναροί σε κάτι άλλο. Και για μένα και για τον κύριο Μπαρνιέ. Μια τέτοια συμφωνία είναι απαραίτητη ε, προϋπόθεση για να υπάρξει συμφωνία ελευθέρου εμπορίου. Θα ήθελα αυτό να είναι πολύ ξεκάθαρο στη διαπραγματευτική εντολή του Συμβουλίου και χαίρομαι που το ψήφισμα αυτό στην παράγραφο 24 συνδέει την αλία οπωσδήποτε με τη γενικότερη συμφωνία. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye και ε, έχουν ζητήσει το λόγο 11 συνάδελφοι. Κλείνει ο κατάλογος, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσουν να μιλήσουν όλοι για ένα λεπτό. Ο κύριος Λόπεθ Αγγιλάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπαρνιέ, κύριε Διαπραγματευτά, τρία χρόνια αγωνιούσαμε για να ε, γλιτώσουμε το άκτακτο Brexit και τώρα έχουμε δέκα μήνες με ένα εξίσου αγωνιώδες ε, και αγχωτικό συνέδριο. Ε, σενάριο μάλλον. Ε, αμοιβαιότητα χρειαζόμαστε και σεβασμό των ε, ευρωπαϊκών προτύπων. Ποτέ δεν ήταν εύκολη η σχέση μας με το Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμα και όταν ήταν μέλος, πόσο μάλλον τώρα που είναι τρίτη χώρα. Δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί φορολογικός παράδεισος μπροστά στην πόρτα μας ή το Γιβραλτάρ να σταματήσει αυτή η παράδοση ε, λαθρεμπορίου, ξεπλήματος και παρανόμων συναλλαγών. Θα πρέπει Επίσης, η κυκλοφορία των πολιτών είναι δεδομένη, η συνεργασία αστυνομική και δικαστική και η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Να μην ξαναυπάρξει ποτέ τέτοιο σκάνδαλο όπως η παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων στο σύστημα πληροφόρηση Σέγγεν, αυτό το σκάνδαλο. Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε μεγάλη προσοχή στην κυκλοφορία των προσώπων και των ελευθεριών. Όλα αυτά τα λέω ως Πρόεδρος Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η κυρία Μαγκίνες, παρακαλώ. Thank Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Μπαρνιέ, χρησιμοποιώ τη δική σας τη φράση Περνάει ο χρόνο, χτυπάει το ρολόι και ξέρουμε ότι χρειάστηκαν δύο-τρία χρόνια προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία αποχώρηση που έχει δύο-τρία ουσιαστικά ουσιαστικά σημεία. Του επόμενου μήνε πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα και να προσέξουμε τι λεπτομέρειε. Το είπαν και οι συνάδελφοι. Ισοτιμία στι σχέσει, θετικέ σχέσει με τον Μένο Βασίλειο και εγώ αυτό εύχομαι στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων αυτών. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρετε ότι οι γενικέ εκλογέ έλαβαν χώρα στην Ιρλανδία και ότι θα έχουμε νέα κυβέρνηση και ελπίζουμε ότι η νέα αυτή κυβέρνηση προσέγγιση θα συνταχθεί, θα αναλάβει την εξουσία το συντομότερο δυνατό, γιατί πολλή δουλειά πρέπει να γίνει. Και ελπίζω ότι θα καταφέρουν να βασιστούν στην καταπληκτική εργασία που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργό, καθώ επίση και η Χέλε Μακιντή, Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, που συνεργάστηκαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε στη συμφωνία αυτή αποχώρηση και ιδίω στο περίφημο Ιρλανδικό Πρωτόκολλο. Οι δέκα μήνε είναι πολύ λίγοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ με την ηγεσία του Ντέβιτ Μακάλαστερ και από κοινού θα πρέπει να συνεργαστούμε για να διατηρήσουμε την ενότητά μα. Ευχαριστώ. Επόμενο ομιλητής είναι ο κύριο Βάλλα. Βάλλα. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε το Ηνωμένο Βασίλειο να γίνει φορολογικός παράδεισος. Ωραία. Η Ποσαχάρια Αφρική κάθε χρόνο χάνει περισσότερα κεφάλαια από όσο παίρνει επενδύσεις και δάνεια νομικά, νόμιμα και παράνομα δρούν οι τράπεζες ε, στο σίτι του Λονδίνου. Μα είναι ήδη φορολογικός παράδεισος. Θέλω να καταλάβω το σκεπτικό σας. Το αθέμητο εμπόριο. Ποιο είναι το ελεύθερο εμπόριο. Θα πρέπει να λέμε τις αλήθειες εδώ. Οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές σκοτώνουν αυτόχθονες λαούς, αγρότες που προσπαθούν να βγάλουν το ψωμί τους Ποιο θα του σταματήσει. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το Brexit ως ευκαιρία να προχωρήσουμε προς ένα σύστημα όπου ο καπιταλισμός ε, δουλεύει στις τοπικές κοινωνίες και δεν κυκλοφορεί σε όλο τον πλανήτη καταστρέφοντας τον κόσμο και τον πλανήτη. Από σοσιαλιστές και δημοκράτες, ε, ο επόμενος ομιλητής, Νεκρέσκο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Προφανώς θα πρέπει να έχουμε θετική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, όχι μόνο υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για το καλό του ίδιου του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τα δεδομένα των πολιτών και στις δύο όχθες της μάχης, θα πρέπει να προστατεύσουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, το είπαν αυτό και συνάδελφοι, αλλά θα πρέπει να έχουμε μια εταιρική σχέση που να περιλαμβάνει και άλλες διαστάσεις, ασφάλεια, άμυνα, προστασία των ε, δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και γιατί όχι η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και σε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα τον θέλουν αυτοί, αν το θέλουμε βέβαια και εμείς. Είμαι πεπισμένο ότι ο κύριο Μπαρνιέ μπορεί πραγματικά να φέρει πέρα με επιτυχία τα καθήκοντα αυτά. Το είδαμε αυτό και στο παρελθόν και κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια στρατηγική εταιρική σχέση, το συντομότερο δυνατό, προκειμένου όλοι αυτοί οι τομεί να προστατεύονται. Σα ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, ο κύριος ε, ε, Τόματς. Microphone. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Thank you, Madam President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μισελ Μπαρνιέ, η κατάσταση σήμερα είναι κάτι το οποίο δεν θελήσαμε εμείς. Εμείς δεν θέλαμε να φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και δεν θέλαμε να βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση που καλούμαστε τώρα να διαχειριστούμε. Τώρα τι να κάνουμε όμως. Ε, σας παρακαλώ να απορρίψετε στεναρά οποιουσδήποτε απαράδεκτους όρους θέσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Διάφορα παράλογα που μπορεί να μας ε, υποβάλουν. Τρία είναι τα σημαντικά για μένα. Σκεφτείτε πρώτον τους Βρετανούς που ήταν κατά του Brexit όταν θα συζητάτε με το Λονδίνο. Δεύτερον, σκεφτείτε ότι έχουμε περίπου 5 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες και πάνω από ένα εκατομμύριο Βρετανούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να τους προστατεύουμε. Και τρίτον, σκεφτείτε ότι η κοινή μας δράση θα πρέπει να ειδωθεί πρόπτικα γιατί κάποια μέρα θα μας ξαναχτυπήσει την πόρτα το Ηνωμένο Βασίλειο. Από το ECR, τα παρακαλώ τώρα. Bogdan. Ε, ε, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Στην Πολωνία λέμε ότι από κοινού μόνο μπορούμε να πετυχαίνουμε θετικά αποτελέσματα. Μόνο μέσω της συνεργασίας επιτυγχάνεται κάτι τέτοιο. Ακριβώς η αρχή αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί και στι διαπραγματεύσει που θα έχουμε με το Μένο Βασίλειο μετά το Brexit. Ένα ερώτημα λοιπόν θέλω να απευθύνω προ τον Επίτροπο. Ξέρετε ότι το Brexit δεν έγινε προκειμένου να διατηρηθεί το εφιστάμενο καθεστώ του status quo. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να συνεργαστούμε, να συμπορευθούμε. Θα πρέπει από κοινού να ταινίσουμε το μέλλον. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο με ενδιαφέρει και εμένα αλλά και του Ευρωπαίου πολίτε. Το ζήτημα τη ασφάλεια. Επ' αυτού θα μπορούσατε κύριε Μπαρνιέ να μα δώσετε περισσότερε λεπτομέρειε. Και έχω κατά νου αυτή τη στιγμή κυρίω την εσωτερική ασφάλεια. Πιστεύετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένε απειλέ στον τομέα αυτό, τι οποίε πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Ντέιλι από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως Ιρλανδή πολίτης πρέπει να πω ότι είχαμε πολύ στενή ε, ιστορία με το Ηνωμένο Βασίλειο και άρρηκτα συνδεδεμένη, όχι πάντα ευτυχία, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό και είναι προς το συμφέρον μας να είναι συνεργασία. Η κυρία Φόντερ Λάιεν μίλησε ε, για ε, κανόνες και για δικαιοσύνη στις επιχειρήσεις. Δικαιοσύνη για ποιον όμως. Αν συνεχίσουν οι κανόνες να ευνοούν τις μεγάλες πολυεθνικές, την βιομηχανία όπλων και τις μεγάλες γεωργικές επιχειρήσεις, οι πολίτες θα μείνουν στην άκρη. Γι' αυτό ο πανίσχυρος ε, Λέο Βαράτκαρ την πάτησε στις εκλογές αυτή την εβδομάδα. Αυτή ήταν η απάντηση του Ιρλανδικού λαού στο νέο φιλελευθερισμό. Έχετε πολλή δουλειά να κάνετε. Κοιτάξτε τι γίνεται με τους γιατρούς ε, και ε, χρειάζεται διοργανική συνεργασία. Συμφωνώ με τους συναδέλφους για τα άλλα ζητήματα και τις παραβιάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά παρακαλώ να μην υποχωρήσουμε στη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Στη συνέχεια. Κύριε Μπαρνιέ, κυρία Πρόεδρε, Μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου βλέπω ότι αρχίζουμε σιγά σιγά και έχουμε κάποια προβλήματα. Ήδη διαφαίνονται αυτά, προβλήματα τα οποία ουσιαστικά θα έχουν να κάνουν με τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Τα ζητήματα όμως αυτά θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να έχουν αρνητική επίπτωση στην μελλοντική εργασία που θα κάνουμε για ένα κοινό πλαίσιο εξωτερική πολιτική και άμυνα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία που έχουμε με τον Ηνωμένο Βασίλειο στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η μόνη εγγύηση που έχουν οι Ευρωπαίοι για μια παγκόσμια ασφάλεια. Θα πρέπει να καταφέρουμε λοιπόν να συντονίσουμε τη σχέση που θα έχουμε με τον Νομένο Βασίλειο στον τομέα επίση τη εξωτερική πολιτική και πιο συγκεκριμένα θεωρώ ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην επίλυση ε, διενέξεων, διενέξεων παγωμένων ή ενεξελίξη στην Συρία, στο Ιράκ. Θα πρέπει από κοινού να αντιμετωπίσουμε τις απειλές τρομοκρατίας. Η περίοδος μετά το Brexit καταδεικνύει αυτή τη στιγμή ότι διανοίγονται νέες ευκαιρίες για μια πιο θετική και στενή συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΗΠΑ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Χάισερ. Ευχαριστώ πολύ. Συζητούμε σήμερα τις μελλοντικές μας σχέσεις με, την, με το Ηνωμένο Βασίλειο. Βεβαίω θέλουμε να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο σχέσεων και όχι απλά μια εμπορική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αυτών λοιπόν θα πρέπει να αποτελέσουμε αξιόπιστου εταίρου που θα μπορούν να δείχνουν εμπιστοσύνη ο ένα στον άλλον όσον αφορά τι προτεραιότητε. Θέλουμε θεμητό ανταγωνισμό, όχι dumping, για να μπορούμε πραγματικά να έχουμε εμπορικέ συναλλαγέ χωρί φραγμούς αυτό όμως σημαίνει ότι και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα επιτρέπεται να δίνει κρατικές ενισχύσεις στις επιχειρήσεις του, ούτε θα μπορεί να αποκλίνει από κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε διευρυμένα δικαιώματα, να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα των πολιτών μας που φοιτούν ή δραστηριοποιούνται οικονομικά στο Ηνωμένο Βασίλειο και να διατηρηθεί το επίπεδο ε, διαβίωσής τους. Ο κύριος Μισελ Μπάνια, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, κύριε Υπουργέ. Με την ευκαιρία της τελευταίας συνόδου στις Βρυξέλλες η ε, Ούρσουλα Φοντελάιεν αναφέρθηκε στον, στη συναισθηματικά φορτισμένη αυτή συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της οποίας αποχαιρετήσατε τους ε, Βρετανούς συναδέλφους ευρωβουλευτές. Θα ήθελα εγώ να καλωσορίσω τώρα τους νέους ευρωβουλευτές που έρχονται να πάρουν τη θέση τους και να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βρίσκεται στο πλευρό τους κατά τη διάρκεια της εντολής τους. Να σε ευχαριστήσω καταρχάς για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε, η οποία μας συγκινεί, αλλά μας ενθαρρύνει παράλληλα και εμένα και όλη την εξαιρετική αυτή ομάδα που με πλαισιώνει. Αναφέρομαι στην ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι και η δική σας διαπραγματευτική ομάδα. Να σε ευχαριστήσω επίσης για το σημαντικό αυτό περιεχόμενο του σχεδίου ψηφίσματός σας που αναφέρεται σε αρχές, που αναφέρεται σε πραγματικές αξίες, που αναφέρεται σε πραγματική τοποθέτηση. Ο διαπραγματευτής σας, ο υποφαινόμενος, πραγματικά τους επόμενους μήνες θα έχω ανάγκη αυτή την αποφασιστικότητα τη δική σας. Τη δική σας τη δέσμευση και την προσήλεση προκειμένου να φέρω εις πέρας τις δύσκολες αυτές διαπραγματεύσεις. Πριν από λίγο η Μέρη Μαγκίνες είπε ότι περνάει ο χρόνος. Ως προς αυτό ως προς το διαθέσιμο χρόνο δηλαδή, να σας πω ότι ο χρόνος αυτής της μεταβατικής περίοδου που προβλέπεται στο πλαίσιο της συμφωνίας αποχώρησης είναι ένας χρόνος όντως πεπερασμένος, περιορισμένος, που θα μπορούσε να επεκταθεί για ένα-δύο χρόνια μέσω μιας κοινή συμφωνίας. Αν δεν επεκταθεί όμως η περίοδος αυτή, τότε το ΜΕΝΟ Βασίλειο θα εγκαταλείψει στις 31 Δεκεμβρίου του 2020 την ενιαία αγορά και την τελωνιακή μας ένωση. Πρόκειται για μία επιλογή, η επιλογή αυτή του χρονιτογράμματος που έχει κάνει ο ίδιος ο Βρετανός Πρωθυπουργός, όχι εμείς οι Ευρωπαίοι. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να καταλάβουμε ότι οι χρονικοί αυτοί περιορισμοί προτού εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο την ενιαία αγορά και την Τελωνιακή Ένωση είναι κάτι το οποίο θα έχει επιπτώσεις και βέβαια την επιλογή αυτή επαναλαμβάνω την έκανε η Βρετανική κυβέρνηση και βέβαια θα πρέπει να να αναλάβουμε την ευθύνη των επιπτώσεων αυτών. Σε καμία περίπτωση εμείς δεν επιλέξαμε αυτό το πολύ στενό χρονοδιάγραμμα. Αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε στο πλαίσιο των συνηθισμένων εμποριακών διαπραγματεύσεων. Ξέρετε ότι όταν διαπραγματευόμαστε, για παράδειγμα, με τον Καναδά ή με την Ιαπωνία, προσπαθούμε να συγκλίνουμε τη θέση μας, να έρθουμε πιο κοντά. Ορισμένοι θεωρούν ότι η σύγκληση αυτή δεν είναι ακόμα επαρκή, αλλά αγωνιζόμαστε για να έρθουμε πιο κοντά. Και αν δεν καταλήξουμε τελικά σε μια συμφωνία με τις χώρες αυτές, δίνουμε στον εαυτό μας περισσότερο χρόνο. Επιτρέπουμε ένα-δύο παραπάνω χρόνια. Στο Καναδά δώσαμε και 7 χρόνια τελικά για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Και στο διάμεσο διάστημα ισχύει το status quo, το εφιστέμενο καθεστώς και για τις δύο συμβαλόμενες πλευρές. Σε συγκεκριμένη όμως περίπτωση, αγαπητοί ευρωβουλευτές, δεν μπορεί να ισχύσει το status quo. Αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία στις 31 Δεκεμβρίου όσον αφορά το εμπόριο, δεν μπορεί να λειτουργήσει το εφιστάμενο καθεστώς. Γιατί καθότι επέλεξε ο Βρετανός Πρωθυπουργό τη μερομηνία αυτή, στις 31 Δεκεμβρίου είχε αποφασιστεί ότι το Μένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Τελειωνιακή Ένωση και την ενιαία αγορά. Και ουσιαστικά θα επιστρέψει κατά αυτόν τον τρόπο, θα μπιστοδρομήσει αν θέλετε, στους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Δηλαδή, πέρα από τους κανόνες που ούτως ή θα κάναμε λόγω του Brexit για όλα τα προϊόντα τα οποία θα έρθουν από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέ... όπω ελέγχουμε ουσιαστικά και όλα τα προϊόντα τα οποία έρχονται από τρίτες χώρες προς την εσωτερική αγορά. Και το κάνουμε αυτό για να προστατεύσουμε πολίτες και επιχειρήσεις. Πέρα λοιπόν από τους ελέγχους αυτούς που ούτως ή άλλως ήταν αγκαίοι, σε συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, αν δεν καταλήξουμε συμφωνία στα τέλη Δεκεμβρίου, θα έχουμε και ποσοστώσεις και τελουνιακούς δασμούς για όλα τα βρετανικά προϊόντα. Να λοιπόν ποια θα είναι η πρώτη και σημαντική επίπτωση, αν δεν καταφέρουμε τελικά να καταλήξουμε σε μια συμφωνία στο περιορισμένο αυτό χρονικό διάστημα που επέλεξε ο Βρετανός Πρωθυπουργό. Κυρίες και κύριοι, κυρία Πρόεδρε, όλες οι πολιτικές ομάδες ζήτησαν να προσιλωθούμε σε ένα υψηλό βαθμό, βαθμό φιλοδοξίας, έχοντας κατά νου την κοινή ιστορία που έχουμε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένο Βασίλειο. Και το λαμβάνω αυτό υπόψη, ιδίω λαμβάνοντας υπόψη τις σκοτεινές σελίδες της ιστορίας του τελευταίου αιώνα. Μόνο και μόνο γεωγραφικά αλλά και από σταρικής πλευράς είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπε ο κ. Λαμπέρτς, να αποτιμήσουμε όλες τις προκλήσεις ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής, περιβαλλοντικές προκλήσεις. Είναι πολύ σημαντικό όμως να είμαστε απόλυτα διαυγείς και σαφείς κάθε φορά που αφουγκραζόμαστε αυτά που έχει να πει η Βρετανική πλευρά και ιδίω ορισμένες δηλώσεις που γίνονται για μια υποθετική χρήση των νέων αυτών δυνατοτήτων που δίνονται στο Ευρωμένο Βασίλειο για να αποκλίνει περισσότερο από τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Brexit. Η ισχυρή λοιπόν φιλόδοξη αυτή η ξεκάθαρη διαυγή σχέση που θέλουμε είναι ακριβώς αυτό το οποίο προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το είπε και η πρόεδρος Φόντερ Λάιν πριν από λίγο. Και αυτό ακριβώς περιλαμβάνεται στην προτινόμενη εντολή για διαπραγματεύσεις, την οποία έχετε ενώπιόν σας και η οποία συζητείται στο Συμβούλιο και ελπίζω ότι θα εγκριθεί στις 25 Φεβρουαρίου. Οι διαπραγματεύσει κυρίες και κύριοι με έναν εταίρο και εδώ πέρα αναφέρομαι σε αυτό που ο κύριος Μπάρι Άντρους πριν από λίγο είναι διαπραγματεύσει με έναν εταίρο ο οποίο θα πρέπει να καταλάβει, και το λέω αυτό με απόλυτη αυστηρότητα και Μία, ότι το άνοιγμα των δικό μας των αγορών, η πρόσβαση στα δεδομένα, κυρία Ένιβελτ, αναφερθήκατε και εσεί αυτό, Απαντώ κύριε Νιβέλτα αυτή τη στιγμή στην ερώτησή σα. Οι ισοδυναμίε όσον αφορά τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε, η Ντανούτα Χούμπνερ αναφέρθηκε σε αυτό, Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι το άνοιγμα το δικό μα των αγορών, η πρόσβαση στα δεδομένα, οι ισοδυναμίε, ή οι ισοδυναμίες στον όσον αφορά τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε θα είναι αναλογικέ σε σχέση με τι κοινέ δεσμεύσει που θα αναλάβουμε προκειμένου να έχουμε ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού, να έχουμε ε, συνέπεια και ομοιομορφία όσον αφορά τους κανονισμούς, όσον αφορά τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε επίσης και την ανάγκη χρηματοπιστωτικής σταθερότητας τη Ευρωπαϊκή Υπήρου και ιδιαίτερα τη Ευρωζώνη. Πολύ γρήγορα να απαντήσω σε κάποιε παρατηρήσει και ερωτήσει. Ο κύριο Μπουρζουά πριν από λίγο αναφέρθηκε στο ζήτημα τη συνεργασία όσον αφορά τη Μαύρη Θάλασσα και τον τομέα τη ενέργεια. Τη Βόρεια Θάλασσα, με συγχωρείτε, στον τομέα τη ενέργεια. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Μπουρζουά, προφανώ να έχουμε μια συνεργασία στην Βόρεια Θάλασσα όσον αφορά τον τομέα τη ενέργειας και αυτό μάλιστα προβλέπεται στο σχέδιο διαπραγματεύσεων αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτόματα, μηχανικά αν θέλετε, υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις από το Brexit. Δεν συμμετέχουν πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι Βρετανοί, άρα θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το πλαίσιο συνεργασίας. Επέλεξε το Ηνωμένο Βασίλειο να μην συμμετέχει στους, στο κοινό αυτό πλαίσιο συνεργασίας, αλλά θα πρέπει να βρούμε ένα διαφορετικό τρόπο συνεργασίας. Ο κύριος Ρανζέλ, πριν από λίγο, και ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ, και πριν από λίγο ο κύριο Τοντσά αναφέρθηκαν στο ζήτημα τη ασφάλεια, εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια. Και αυτό περιλαμβάνεται στην προτινόμενη εντολή διαπραγματεύσεων. Προβλέπονται πολλέ διαπραγματεύσει στον τομέα τη εσωτερική ασφάλεια, συνεργασία όσον αφορά τι απελάσει, συνεργασία με την Eurojust, την Europol, καταπολέμηση τη παράνομη, ε, τη νομοποίηση παράνομων εσόδων, η Σύμβαση Προύν και πολλοί άλλοι μηχανισμοί προβλέπονται όσον αφορά την προστασία των πολιτών. Ο κύριος Αλεξανδρόφ πριν από λίγο επίσης αναφέρθηκε και στην εξωτερική ασφάλεια ως προς αυτό και αναφερόμενος ιδιαίτερα στην άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Θα ήθελα να σας πω ότι το Brexit λογικά δεν θα πρέπει να έχει επιπτώσει όσον αφορά τη διμερή συνεργασία που πολλές από τις δικές σας χώρες ήδη έχουν με το Μένο Βασίλειο. Αναφέρομαι σε ομονωμένη διμερή συνεργασία και βέβαια δεν θα πρέπει να έχει και επιπτώσεις αυτό που κάνουμε από κοινού στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Στα πλαίσια των διαπραγματεύσεών μα, αναφερόμαστε στη συνεργασία που θα έχουμε μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και του Βασιλείου, ιδίω σε διάφορε νέε πρωτοβουλίε στον τομέα τη άμυνα. Εμεί ε, θέλουμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσει και για το άτομα αυτό, το αίτημα, το τομέα αυτό, με συγχωρείτε. Η πολιτική διακήρυξη αναφέρεται επίση και στην άμυνα και στην εξωτερική πολιτική και θα έλεγα ότι χρειαζόμαστε ένα συγκεκριμένο κείμενο για τους τομείς αυτούς προκειμένου στα νομικά κείμενα που θα προκύψουν να προβλέπεται μια διοικητική ή πολιτική συνεργασία, για παράδειγμα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας ή αν θέλετε για την καταπολέμηση των κυβερνοεπιθέσεων ή για την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα των μυστικών πληροφοριών ή για να μπορούν οι Βρετανοί, εφόσον το θέλουν, να συμμετέχουν σε εξωτερικέ αποστολέ, στρατιωτικέ ή μη στρατιωτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αναφέρομαι βέβαια και στην πολιτική συνεργασία με μια χώρα η οποία είναι πολύ σημαντική και παραμένει μόνιμο μέλο του Συμβουλίου Ασφαλεία των Ηνωμένων Εθνών. Όλα αυτά τα κείμενα διαπραγματεύσεων μπορούμε να τα συζητήσουμε περαιτέρω. Θα πρέπει να εμπλέκονται και τα δύο συμβαλόμενα ένα μέρη. Εμεί παραμένουμε ανοιχτοί και διαλλακτικοί προκειμένου να καταφέρουμε να βελτιώσουμε την κοινή διαχείριση της σταθερότητας της Υπήρου μα. Επίσης, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Πριν από λίγο, κυρία Τέρη Ράνκιν αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Εράσμου, μα προφανώς και θα πρέπει να συνεχίσουμε την συνεργασία, την πανεπιστημιακή, τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας, τη συμμετοχή των Βρετανών εφόσον το επιθυμούν στα ευρωπαϊκά προγράμματα και θα προβλεφθούν και συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις ήδη από το Μάρτιο για το σύνολο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος Εράσμους, αλλά και εκεί πέρα πάλι θα έχουμε ένα οικονομικό πλαίσιο και ένα πλαίσιο διαχείριση διαφορετικό από το σημερινό. Η κυρία Ντανούτα Χούμπνερ αναφέρθηκε πριν από λίγο στι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε και τη σχέση που θα πρέπει να έχουμε στον τομέα αυτό με το Ηνωμένο Βασίλειο. Πέρα από οτιδήποτε αυτή τη στιγμή προβλέπεται στην προτινόμενη εντολή διαπραγματεύσει και πέρα από αυτά τα οποία συνήθω κάνουμε στι συμφωνίε με τι τρίτε χώρε, δεν προβλέπονται συγκεκριμένε διαπραγματεύσει όσον αφορά τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε. Από την άλλη, θα πρέπει να έχουμε μια κάποια σχέση στον τομέα αυτό με το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω τη ιδιαίτερη θέση που έχει το Λονδίνο και ιδιαίτερα το ΣΥΤΙ στον τομέα αυτό και η Ντανούτα αναφέρθηκε πριν από λίγο στις ισοδυναμίες στην εργαλειοθήκη αυτή που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε, αν θέλετε, λοιπόν, την εργαλειοθήκη αυτή των ισοδυναμιών. Δεν διαπραγματευόμαστε όμως γι' αυτό με το Ηνωμένο Βασίλειο. Προσπαθούμε να επαληθεύσουμε πώ έχουν τα πράγματα και όταν το κρίνουμε αναγκαίο τότε μπορούμε να προβλέψουμε συγκεκριμένε ισοδυναμίε και συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικούς τομείς. Αυτό κάναμε με τον Καναδά, αυτό κάνουμε με τις ΗΠΑ, στην Ιαπωνία και το σύστημα αυτό λειτουργεί θετικά. Για ποιο λόγο λοιπόν να μην λειτουργήσει αποτελεσματικά και με το Ηνωμένο Εποφελούμε επίση ευκαιρία για να πω προ ορισμένου Βρετανού αξιωματούχου ότι θα πρέπει να υπάρχει καμία ψευδέστηση ω προ το ζήτημα αυτό. Δεν πρόκειται να προβλεφθεί μια γενική σφαιρική ισοδυναμία όσον αφορά τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε και δεν πρόκειται να υπάρχει συνδιαχείριση οικονομικών ισοδυναμιών με την Ηνωμένο Θα διατηρήσουμε εμεί την χρησιμοποίηση των εργαλείων αυτών και θα έχουμε απόλυτη αυτονομία στις αποφάσεις που θα λάβουμε. Και ξεχνάμε ότι ε, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που μας κάνουν να πρέπει να αναλάβουμε δράση στον τομέα αυτό τη στιγμή που εμείς επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και της ε, Ένωσης Κεφαλογικών Αγορών. Όσον αφορά την Αλία και αναφέρομαι αυτή τη στιγμή στον κύριο Μπελαμή, στον κύριο Πέτερ, στην κυρία Σκανταλμόζε, στον κύριο, στην κυρία Αγγιλέρα που αναφέρθηκαν στον τομέα της Αλίας. Ένα τομέα τον οποίο το γνωρίζω πολύ καλά γιατί είχα την τιμή να είμαι και Υπουργό Αλία για κάποια χρόνια στη δική μου τη χώρα, τη Γαλλία. Ω προ τον τομέα τη Αλία, λοιπόν, να σα πω ότι η αμοιβαία πρόσβαση στα ύδατα και στις αγορές, αμοιβαία πρόσβαση στα ύδατα και από τις δύο πλευρές και στις αγορές και από τις δύο πλευρές αποτελεί ένα τμήμα της, αναπόσπαστο τμήμα της εμπορικής συμφωνίας και αναπόσπαστο τμήμα του ισότιμου πεδίου ανταγωνισμού που θέλουμε να έχουμε στα πλαίσια διαπραγματεύσεων. Κυρίες και κύριοι, εμείς ε, ανέκαθεν σεβόμασταν όλον ότι λυπούμεθα για αυτή την επιλογή των ε, Βρετανών πολιτών να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πρωθυπουργό Μπόρι Τζόνσον, τον οποίο σεβόμαστε, είπε ότι αποχωρώντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αποχωρεί από την Ευρώπη και εμεί χαιρόμαστε γι' αυτό. Το ζήτημα όμω το οποίο τίθεται αυτή τη στιγμή και το οποίο δεν μα έχει δοθεί μια απάντηση είναι πολύ απλό αλλά πολύ σοβαρό. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποχωρεί από την Ελληνική Ένωση και την ενιαία αγορά. Θέλουν όμω να αποχωρήσουν, να απομακρυνθούν από το οικονομικό, κοινωνικό μα μοντέλο, το ρυθμισμένο αυτό μοντέλο που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά γιατί από κοινού το οικοδομήσαμε εδώ και 47 χρόνια. Αυτό είναι το ερώτημα επί του οποίου περιμένουμε μια απάντηση. Ποια απόσταση τελικά θέλει να έχει από εμά το Ηνωμένο Βασίλειο, πόσο θέλει να απομακρυνθεί από το δικό μας οικονομικό, κοινωνικό και ρυθμιστικό μοντέλο. Και πρέπει να σας πω και το λέω αυτό με απόλυτη σαφήνεια και νυφαλιότητα, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αυτό το οποίο θα θέσει το επίπεδο φιλοδοξία που θέλει για τι μελλοντικέ σχέσει μαζί μα. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αυτό το οποίο θα επιλέξει το επίπεδο ρυθμιστική συνέπεια, το οποίο θα κρίνει τελικά και το επίπεδο φιλοδοξίες που θα έχουμε, το μέλλον Βασίλειο είναι αυτό το οποίο θα αποφασίσει και το επίπεδο του ανταγωνισμού που θέλει να έχει μαζί μας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να προβληματιστεί το Μένο Βασίλειο προς το ερώτημα αυτό που έθεσα. Και να κάνω και τρει ακόμα πολύ σύντομε σκέψει. Κυρίε και κύριοι, πάντα έλεγα την αλήθεια ενώπιον σα και αυτό θα συνεχίζω να κάνω. Το Brexit δεν μπορεί να είναι business as usual. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με την πεπατημένη. Έχουμε αλλαγέ σε όλου του τομεί. Ορισμένε αλλαγέ και τροποποιήσει μπορεί να είναι μικρέ και προσωρινέ, άλλε θα είναι μεγάλε και καθοριστικέ. Το Ηνωμένο Βασίλειο ουσιαστικά κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο να χάνει το λεγόμενο χρηματοπιστωτικό διαβατήριο. Δεν θα υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση. Λόγω του Brexit, σε κάθε περίπτωση, από την 1η Ιανουαρίου του 2020 θα πρέπει να επιβάλλουμε ελέγχου σε όλα τα προϊόντα τα οποία θα εισέρχονται στην εσωτερική μα αγορά, όπω κάνουμε για οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα. Την προστασία αυτή την οφείλουμε στου δημόσιου προπολογισμού μα, στον ενωσιακό προπολογισμό, στι επιχειρήσει μα και στου πολίτε μα. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε business as usual, αλλά θα πρέπει να περιορίσουμε και τι αρνητικέ επιπτώσει. Αυτό το προβλέπουμε σε κάθε συμφωνία. Δεύτερον, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να τηρήσουμε τη συμφωνία αποχώρησης. Δεν πρόκειται για κάτι το αμεληταίο. Είναι μια συμφωνία 600 σελίδων την οποία επικυρώσατε και εσείς αλλά και η Βουλή των Κοινοτήτων θα πρέπει λοιπόν να εφαρμοστεί. Επομένω, δημοσίω μπροστά σα και ενώπιον του Συμβουλίου θα έρχομαι να μιλάω για την προπαρασκευαστική αυτή περίοδο κατά τη διάρκεια του 2020 και θα, θα αναφέρομαι στο πώ εφαρμόζεται η συμφωνία αυτή και όλου ιδιαίτερο στο πρωτόκολλο τη Ιρλανδία για την προάσπιση αυτή τη έφθραστη ειρήνη. Οι διαπραγματεύσει θα είναι δύσκολε, πολύ δύσκολε, κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, όλα τα σενάρια και τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, ακόμα και το να μην καταλήξουμε τελικά σε μια συμφωνία στις 31 Δεκεμβρίου του 2020. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια στα πλαίσια απόλυτη εμπιστοσύνη και σεβασμού με απόλυτη νεφαλαιότητα να προωθήσουμε τι διαπραγματεύσει αυτέ. Πέρα από τι καθημερινέ δυσκολίε διαπραγμάτευση, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πάντα την απόλυτη προοπτική να καταλήξουμε σε μια φιλόδοξη συμφωνία εξ ονόματό σα με μια χώρα η οποία θα είναι πάντα φίλο και εταίρο Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, επαναλαμβάνω την απόλυτη προσήλωσή μου να προασπίσω την ακαιρεότητα της εσωτερικής μας αγοράς συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων την ακαιρεότητα μιας εσωτερικής αγοράς που ποτέ δεν θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μπορεί να είστε σίγουροι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η διαπραγματευτή σα, ο υποφαινόμενο, θα είμαι πάντα στο πλευρό σα, πάντα θα σα ακούω, θα είμαι πάντοτε στη διάθεσή σα και όπω το έλεγα όλα αυτά τα τρία χρόνια, και όπω το είπα και απέναντι στην ομάδα επικεφαλή τη οποία ήταν ο κύριο Φερχόφστατ στο παρελθόν και τώρα ο κύριο Μακάλιστερ αναφέρομαι στην ομάδα συντονισμού και ενώπιον όλων των προέδρων των πολιτικών ομάδων επαναλαμβάνω τη διαθεσιμότητά μου για να βρίσκουμε πάντα στο πλευρό σα και να συνεργάζομαι μαζί σα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να κλείσει τη συζήτηση το λόγο έχει το Συμβούλιο. Παρακαλώ, Υπουργέ. Ευχαριστώ συνάδελφοι και εγώ να χαιρετήσω τα νέα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου και προσβλέπω στις συζητήσεις που θα έχουμε. Με την ψηφοφορία σας για το ψήφισμα για την εντολή διαπραγμάτευσης για τη νέα σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο θα τροφοδοτήσετε με ε, έγκαιρο τρόπο την ε, στάση μας. Πρέπει να οικοδομήσουμε μία σχέση η οποία θα είναι αμοιβαία, θα ε, τηρεί τους ίσως ανταγωνισμού και θα είναι ολοκληρωμένη. Οι μακροσκελείς διαπραγματεύσεις, οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσουν σε διάφορους τομείς, θα χρειαστούν συζήτηση τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Αυτή η νέα φάση βεβαίως δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχάσουμε την συμφωνία αποχώρησης. Πρέπει να επαγρυπνούμε όσον αφορά την εφαρμογή της. Κατά κύριο λόγο όσον αφορά την διατήρηση των δικαιωμάτων των πολιτών, είτε κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου είτε και κατά τη διάρκεια των μελλοντικών μας σχέσεων. Όμως η επαγρύπνηση αυτή θα πρέπει να ε, έχει το βλέμμα της στραμμένο στη δημιουργία μιας νέας οικονομικής ε, σχέσης όπου μέσω της διακυβέρνησης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ενιαία αγορά ε, και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Θέλουμε την συνεργασία σας και σε αυτό το τομέα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται η συζήτηση αυτή. Ε, έχει κατατεθεί ένα σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο θα ψηφιστεί αύριο. Να σας πω επίσης ότι ολοκληρώνουμε τη συζήτηση για αυτό το ημέρι, για οι σοσιαλιστές ε, διαβίβασαν μια, ένα αίτημα για αλλαγή των συντονιστών στις επιτροπές. Ε, από σήμερα ε, καταγράφονται στα πρακτικά αυτά τα αιτήματα και θεωρούνται κεκριμένα. Επόμενο θέμα είναι η, συζήτηση, η κοινή συζήτηση για το Βιετνάμ. Έχουμε τέσσερις εκθέσεις και συστάσεις από τον συνάδελφο Μπουρζουά, ο οποίος και θα λάβει πρώτος τον λόγο. Παρακαλώ για λεπτά. Σας ευχαριστώ αγαπητή Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, αγαπητέ Επίτροπε. Αύριο, συνάδελφοι, θα ψηφίσουμε για την ε, Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών και ε, Συμφωνία Προστασίας Επενδύσεων με το Βιετνάμ. Είναι οι πρώτες τέτοιου είδους συμφωνίες ε, σύγχρονο τύπου που καλείται το Κοινοβούλιο να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μοναδική ευκαιρία για το Κοινοβούλιο να τονίσουμε την φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταστεί ένας γεωπολιτικός πρωταγωνιστής. Όχι ως αυτοκρατορία που επιβάλλει κανόνες, αλλά Ω μια παγκόσμια δύναμη που υπερασπίζεται την πολυμερή συνεργασία, αντιστέκεται απέναντι στους προστατευτισμού και την χείρα βοηθεία σε εταίρου όπω είναι το Βιετνάμ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εναπόκειται να προάγει το εμπόριο που βασίζεται σε κανόνε και να δείξει το παράδειγμα ότι το εμπόριο αποδίδει, ότι το εμπόριο φέρνει του λαού πιο κοντά και ανεβάζει παγκοσμίω τις προδιαγραφέ. Προδιαγραφέ ασφαλεία, ε, εργασία, περιβάλλοντο και ανθρωπίνων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, τίθεται και ένα θέμα αξιοπιστίας. Θα πρέπει να δείξουμε στο Βιετνάμ αλλά και σε μελλοντικού εμπορικού εταίρου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αξιόπιστο εταίρο που τηρεί τις ε, δεσμεύσει τη, Ότι μπορεί ακόμα να διαπραγματεύεται, να υπογράφει και να ολοκληρώνει και να συνάπτει εμπορικέ συμφωνίε. Αγαπητοί συνάδελφοι, οκτώ χρόνια μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Βιετνάμ, το Κοινοβούλιο έχει πλέον την ευκαιρία να συζητήσει την σημαντικότερη και συνολικότερη συμφωνία ε, εμπορικών συναλλαγών με μια χώρα μεσαίου το Πρωτοφανέ στην ιστορία. Είναι ορόσημο για ε, τη δέσμευση και τη συνεργασία της Ευρώπης με αναδυόμενες οικονομίες. Αν κοιτάξουμε αυτή την εμπορική συμφωνία, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε πρώτα απ' όλα την οικονομική αξία που θα δώσει τεράστια όθηση ε, για στην εφημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Βιετνάμ. Είναι καταπληκτική ευκαιρία για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές, για τους εξαγωγείς και τους επενδυτές καταργεί το 99% των δασμών μέσα σε μία επταετία, πράγμα που θα καταλήξει σε επιπλέον εξαγωγές και προς τις δύο κατευθύνσεις. Θα έχουμε ε, δεκάδες χιλιάδες καλύτερες θέσεις εργασίας, πιο ποιοτικέ και κατά μέσο όρο καλύτερα αμοιβόμενες. Θα ε, ανέβουν και παγκόσμιως οι διεθνείς προδιαγραφές. Εδώ μειώνονται και, και οι μη εμπορικοί φραγμοί και το, τα έξοδα για τις εταιρείες μας. Ε, κερδίζουμε καλύτερη πρόσβαση στις αγορές ε, και στις δημόσιες συμβάσεις και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, είναι παλόμενη η βιομηχανία στο Βιετνάμ, η οικονομία, πάνω από 90 εκατομμύρια καταναλωτές, δυναμική μεσαία τάξη και εργαζόμενους νέους και πραγματικά θέλει να ασπαστεί ε, νέους κανόνες και σύγχρονες προδιαγραφές. Ήταν η πρώτη χώρα, ακόμα και πριν τον Καναδά, που ε, δέχτηκε ε, ένα σύστημα λύσεις διαφορών με τους επενδυτές, με ανεξάρτητους δικαστές, με κανόνα δεοντολογίας, με προστασία των δικαιωμάτων και του δικαιώματος να ρυθμίζεις και πιο εύκολη πρόσβαση ε, στα δικαστήρια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η συμφωνία αυτή λοιπόν φέρνει νέες ευκαιρίες για τις εταιρείε και για τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και για τις μικρομεσαίες εταιρείε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το Βιετνάμ είναι και η πύλη προς ολόκληρη την περιοχή ΑΣΕΑΝ. Η συμφωνία αυτή είναι ε, υλοποίηση και η ενσάρκωση του παλιού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για εμπόριο περιφέρεια προς περιφέρεια. Στόχο έχει να προωθήσει και να προστατεύει τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες και τις προδιαγραφές. Το Βιετνάμ ε, σέβεται και έχει σαφείς ε, προθέσεις να ακυρώσει δύο βασικές ακόμα συμβάσεις του ΆΕΛΟ. Αναθεώρησε τον εργατικό κώδικα, βελτιώνει την κατάσταση Τη εργασία και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει την ε, Συμφωνία του Παρισίου για ε, την κλιματική αλλαγή. Για όλους αυτούς τους λόγους και επειδή πρόκειται για δημιουργία ευημερία με ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση να λαμβάνει ευθύνη να θέσει παγκόσμιες προδιαγραφές και να πρωταγωνιστήσει σε ένα εμπόριο που να βασίζεται σε κανόνες ε, σε καιρούς όπου ενδύνονται ε, τα προβλήματα στο εμπόριο και ε, αυξάνεται ο προστατευτισμός. Σα ζητώ να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μας, έτσι ώστε οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο λαός του Βιετνάμ να συσφίξουν περαιτέρω τις σχέσεις τους στο μέλλον, έτσι ώστε να επιτρέψουμε ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο για να φέρουμε πιο κοντά ακόμα τους λαούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Καλωσορίζω τον Επίτροπο κύριο Χόγκαν στην Ομίγυρη, ο οποίος θα λάβει αμέσω το λόγο εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ε, Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, η Συμφωνία Ελευθερών Περίου και η Επενδυτική Συμφωνία με το Βιετνάμ είναι οι πιο φιλόδοξες συμφωνίε που έχουμε ποτέ συνάψει με αναπτυσσόμενη χώρα θα μας επιτρέψουν να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τους εμπορικούς και επενδυτικούς μας δεσμούς και θα μας δώσουν τη δυνατότητα να ενισχύσουμε τη συνεργασία ε, στο πλαίσιο άλλων ευρωπαϊκών μηχανισμών, όπως είναι την άναρχια, όπως είναι η αναρχιαλία. Ακολουθεί το παράδειγμα ε, άλλων συμφωνιών όπως είναι με την Κορέα, το Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη. Και υπάρχει, ε, είναι μια ευκαιρία για να ενισχύσουμε τη σχέση μας με την ε, περιοχή ΑΣΕΑΝ. Είναι μια χώρα με εκατομμύρια καταναλωτές εργαζόμενους και πρέπει να καταργήσουμε τους δασμούς και τις, τα εμπόδια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα αλκοολούχα ποτά, στον μηχανολογικό εξοπλισμό, στα αυτοκίνητα. Με αυτόν τον τρόπο θα άρουμε και ε, εμπόδια για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Για πρώτη φορά ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα μπορούν να συμμετέχουν στις δημόσιες προμήθειες και θα υπάρχουν και πλέον ε, θα υπάρχει προστασία για τα ευρωπαϊκά προϊόντα όσον αφορά την προέλευσή τους και τις ονομασίες προέλευσής τους. Επίσης ε, προβλέπονται ε, κανόνες για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η Συμφωνία Προστασία των Επενδύσεων, που είναι παρόμοια με εκείνη που έχουμε με τον Καναδά και την Σιγκαπούρη, προβλέπει ένα σύγχρονο νέο σύστημα για την προστασία των επενδύσεων με την πρόβλεψη και ενός δικαστηρίου. Όμως υπερβαίνουν οι σχέσεις μας ε, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Θέλουμε, ε, υπάρχει, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο κεφάλαιο που αφορά την